συζήτηση για το θέμα αυτό. Η ψηφοφορία θα λάβει χώρα αύριο στις 11.30 και τώρα φτάνουμε στο τελευταίο θέμα. Πρόκειται για την έκθεση Higgins, στρατηγική για την υπηρεσία τηλεδιοδίων, σύστημα τελών με αυτοκόλλητο για τα ελαφρά οχήματα ΙΧ. Η έκθεσή μου, κύριε Πρόεδρε, σαφώς και θα πρέπει να μας οδηγήσει σε μια βιώσιμη πολιτική υποδομών που θα μας οδηγήσει στο μέλλον. Επίσης θα πρέπει να δούμε πώς η αρχή ορυπαίνων πληρώνει θα πρέπει να εφαρμοστεί στο μέλλον με ένα ηλεκτρονικό σύστημα τηλεδιοδίων στην Ευρώπη. Γνωρίζω ότι αυτό το σύστημα που μέχρι τώρα έχει εφαρμοστεί είναι απογοητευτικό. Είναι απαραίτητο λοιπόν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ξαναδεί με ποιο τρόπο θα μπορούσε να μεταρρυθμίσει την υπάρχουσα νομοθεσία χρησιμοποιώντας ένα αποτελεσματικό σύστημα τηλεδιαδίων. Ένα σύστημα ηλεκτρονικό γιατί από ό,τι είδαμε οι χρήστες αυτών των διοδίων καθώς και οι χειριστές του υπάρχοντος συστήματος θέλουν να βρουν ένα σύστημα που να αντιποκρίνεται στις πραγματικές ανάγκες των χρηστών. Ένα ενιαίο σύστημα το οποίο θα βασίζεται σε πολιτικούς στόχους και όχι τεχνολογικούς. Θα πρέπει να υπάρχει μία μονάδα η οποία να αντιμετωπίζει τις σημερινές ανάγκες και η οποία Μέχρι σήμερα οι αυτοκινητόδρομοι οι οποίοι δεν επιβάλλουν διόδια θα πρέπει να εξοπλιστούν με τον νέο εξοπλισμό και θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αντιμετωπίσει αυτές τις δυνατότητες επιβολής τέλων και διοδίων. Ένα νέο σύστημα θα πρέπει να μας επιτρέψει να συνεχίσουμε να επιβάλλουμε διόδια και τέλη, τα οποία βέβαια θα είναι ανάλογα με τη χρήση των ε, διοδίων. Θα πρέπει να υπάρχουν δυνατότητες πληρωμής ε, μηνιαίων τελών, ε, είτε ημερήσιων, ανάλογα με την συχνότητα χρήσης των διαδρομών και των αυτοκινητοδρόμων θα πρέπει να υπάρχει ε, αυτοκόλλητη ετικέτα η οποία να καθορίζει τα ποσά με μηνιαία τέλη είτε ετήσια τέλη. Και βεβαίως από εδώ και πέρα τα κράτη-μέλη θα έχουν μία δυνατότητα υιοθέτηση των συστημάτων αυτών ανάλογα με την υπάρχουσα υποδομή. Κατά την άποψή μου και κατά την άποψη πολλών κρατών μελών θα πρέπει να στοχεύσουμε μία τέτοια αυτοκόλλητη ετικέτα και βεβαίως θα συνεχίσουν να υπάρχουν κάποιοι δρόμοι χωρίς τέλη, χωρίς διόδια, αλλά σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να υπάρχει μια διακριτική χωρις διοδια αλλα σε καθε περιπτωση θα πρεπει να υπαρχει μια διακριτικη ευχαίρεια των κρατών μελών, αφού προηγουμένως ε, εκφραστούν οι επιθυμίες της Επιτροπής και του Συμβουλίου. Μέχρι αυτή η επιθυμία, αυτό το όνειρο να γίνουν πραγματικότητα. Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Σίγητα. Νομίζω ότι μπορούμε κατευθείαν να προχωρήσουμε στη διαδικασία Catch the Τέσσερις ομιλητές έχουν ζητήσει το λόγο. Μπορούμε να το δώσουμε και στους τέσσερις. Ο κύριος Μπάνκι είναι ο πρώτος. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Πιστεύω ότι όλοι μπορούμε να συμφωνήσουμε πως ε, αυτό το σύστημα που σήμερα υπάρχει στην Ευρώπη δεν λειτουργεί ικανοποιητικά και θα συμφωνήσω εδώ ιδιαίτερα με τον ε, εισηγητή ότι δεν είναι αρκετά αυστηρή η υπάρχουσα νομοθεσία στα κράτη-μέλη, δεν υπάρχουν ε, αρχές οι οποίες να διέπουν όλη την Ευρώπη για τα τέλη, δεν υπάρχει μια ενιαία υποδομή, ένας ενιαίος εξοπλισμός και συμφωνώ απολύτως με τον κύριο Higgins, ο οποίος λέει ότι ο χρήστης θα πρέπει να γνωρίζει τις αρχές και η αρχή ορυπαίνων πληρώνει είναι κάτι που θα πρέπει να επιβληθεί σε όλη την Ευρώπη. Χρειαζόμαστε λοιπόν περαιτέρω επενδύσεις από τις οποίες να μπορούν να υποφεληθούν όλοι οι Ευρωπαίοι πολίτες. Και νομίζω ότι μόνο μια τέτοια νέα λύση θα είναι ικανοποιητική. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δανέλης με την επιβολή τελών χρήσης υποδομών στους αυτοκινητοδρόμους τα κράτη μέλη εφαρμόζουν την αρχή που θέλει τον χρήστη να πληρώνει για τη χρήση του αυτοκινητοδρόμου αντί του φορολογουμένου. η πρακτική αυτή επιτρέπει τον δίκαιο ανταγωνισμό για παράδειγμα στη μεταφορά εμπορευμάτων αφενός μεταξύ των οδικών μεταφορών και αφετέρου των θαλάσσιων και σιδηροδρομικών. η επιβολή των τελών αυτών είναι λοιπόν καταρχήν δικαιολογημένη φτάνει να απορρέει από σωστή τιμολόγηση η οποία να αντανακλά το κόστος κατασκευής και φθοράς τη υποδομή. ωστόσο η έκθεση του συναδέλφου higgins ορθά εκφράζει την απογοήτευσή μας όσον αφορά δύο εμπόδια στη διαμόρφωση ενός σύγχρονου και αποτελεσματικού συστήματος διοδίων στην ευρώπη που πρέπει να αρθούν. πρώτο η ακινησία των κρατών μελών και σχετικών κλάδων όσον αφορά τι διαδικασίε οργάνωσης Ευρωπαϊκή ευρωπαϊκής υπηρεσίας τηλεδιοδίων και δεύτερο η ασυμμετρία που προκαλεί ο τρόπος χρήσης των συστημάτων βινιέτας από αρκετά κράτη μέλη που με έμεσο τρόπο πρημοδοτούν του πολίτε τους έναντι άλλων ευρωπαίων χρηστών. Σας ευχαριστώ. E, Ευχαριστώ. Χαίρομαι πάρα πολύ που επιτέλους δέχτηκε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το νέο ότι το νέο σύστημα 2.2 ήταν αποτυχία μέχρι στιγμής. Τα διάφορα εργαλεία που χρησιμοποίησαν τα κράτη-μέλη για τη χρέωση που λειτουργούν ε, βινιέτα, μικροκύματα, ηλεκτρονικά διόδια, διάφορα διαφορετικά συστήματα, τα οποία όμως δεν έχουν εναρμονιστεί ακόμη ε, νομίζω ότι τα δορυφορικά τηλεδιόδια είναι η λύση του μέλλοντος, γιατί μόνο έτσι μπορούμε να καταμετρήσουμε το χρόνο χρήσης ε, από τον οδηγό και να υπολογίζουμε ε, και το, τη ρήπανση που προκαλεί ο κάθε χρήστης. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό για τους καταναλωτές. Να, πρέπει να προσπαθήσουμε Επίσης για τις μεταφορές ε, να θεσπίσουμε ένα νέο σύστημα, τις μεταφορές εμπορευμάτων ε, και νομίζω ότι η παρακολούθηση της κυκλοφορίας έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για όλους. Ευχαριστούμε και τέλος ο κύριος Φερέιρα. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Οι οδικές υποδομές ε, θα πρέπει να καλύπτουν ε, οικονομικές ανάγκες αλλά και προσωπικές ανάγκες κινητικότητα των ανθρώπων και των εμπορευμάτων. Αυτές οι ανάγκες θα πρέπει να εξεταστούν στο ειδικό περιφερειακό τους πλαίσιο. Θα πρέπει να δούμε πώς λειτουργεί η κάθε υποδομή και για να δούμε αν θα πρέπει να εισαγαγούμε τηλεδιόδια ή όχι και αν πρέπει κανείς να πληρώνει ή όχι. Παραδείγματο χάρη στην Πορτογαλία νέα διόδια στους αυτοκινητοδρόμους όπου δεν υπήρχαν παλαιότερα διόδια είχε καταστροφικά αποτελέσματα για την τοπική οικονομία, για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις, για την κινητικότητα των οδηγών και για την ίδια την υποδομή τους αυτοκινητοδρόμους ε, και ουσιαστικά ε, η χρέωση των ε, δύο δίων ε, χρηματοδοτεί την κατασκευή αυτών, την κατασκευή του νέου συστήματος. Δεν μπορούμε λοιπόν να αγνοήσουμε την καταστροφική και τραγική εμπειρία που είχαν τα κράτη-μέλη που προσπάθησαν να εισαγάγουν τέτοια συστήματα μέχρι στιγμή. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε, λέει ο Πρόεδρος. Η τελευταία παρέμβαση θα είναι αυτή του Επιτρόπου, του κ. Σέμετα. Ευχαριστώ, Πρόεδρε, αξιότιμα μέλη του Κοινοβουλίου. Ευχαριστώ και εγώ τον εισηγητή και όλα τα μέλη για τις πολύ επικοδομητικές ε, παρατηρήσεις τους. Όσον αφορά ένα νέο σύστημα τελών για όλες τις κατηγορίες των χρηστών των ε, αυτοκινητόδρομων, συμφωνούμε ότι αυτή η πρωτοβουλία είναι κάτι που θα πρέπει να εξεταστεί για γιοταχή και χωρίς ε, διακρίσεις ε, κατά των χρηστών, για όλους τους χρήστες δηλαδή των αυτοκινητοδρόμων, θα πρέπει με ευελιξία τα κράτη-μέλη να μπορούν να επιβάλλουν τέλη και διόδια, έτσι ώστε να αποφευθεί συμφόρηση σε κάποιες περιοχές και αυτό είναι κάτι που το βλέπουμε σαν αιτήματα πολλών τροπολογιών. Είναι κάτι που το ζητούν αρκετά κράτη-μέλη. Θεωρούμε πραγματικά ότι η δημιουργία ενός τέτοιου συστήματος τελεδιδιών δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να καταργήσουν από τη μία μέρα στην άλλη τα υπάρχοντα συστήματα. Ο σκοπός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής του Ευρωπαίου Νομοθέτη είναι να διασφαλίσουμε τα περιφερειακά προγράμματα και ολοκληρώνοντας θα ήθελα να πω ότι η συνέχιση των συστημάτων που υπάρχουν θα πρέπει να εξεταστεί πολύ προσεκτικά, καθώς και οι νέες πρωτοβουλίες, νομοθετικές πρωτοβουλίες για την επίτευξη ενός νέου συστήματος. Σας ευχαριστώ πολύ. Ολοκληρώθηκε και η συζήτηση για αυτό το σημείο της ημερήσιας διάταξης. Η ψηφοφορία θα γίνει αύριο στις 11.30. Η επόμενη συνεδρίαση θα λάβει χώρα αύριο το πρωί.